Ε, στην αδειοδότηση ε, τεχνικών γενετικής, ε, η χρήση ζυζανιοκτώνων είναι πράγματα που δεν μπορούμε να αφήνουμε στην απόφαση της Επιτροπής. Δεν μας καθησυχάζει κάτι τέτοιο. Δεν μας καθησυχάζει ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας και άλλες συμπεριφορές ψηφοφορίας τελικά γίνονται ε, είναι σαν να λένε όλοι ναι εντάξει θα κάνουμε ό,τι γίνει αλλά εγώ δεν θέλω να βρέξω τα πόδια μου. Οι αλλαγέ που προτείνονται ε, θεωρούμε ότι είναι θετικέ. Η αλλαγή των μεθόδων, η Επιτροπή ε, Προσφυγών και όλα τα λοιπά. Και την πρόταση που είπαν κάποιοι συνάδελφοι θεωρώ ότι είναι λάθο να αποσυρθεί η πρόταση τη Κομισιόν και να γίνει μια νέα πρόταση που να αρέσει καλύτερα στο Συμβούλιο. Πρέπει να καταλάβουμε σαφώ ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση δεν θα είναι παρά μια αποδυναμωμένη εκδοχή τη σημερινή πρόταση. Τελικά αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσουν οι εργασίες για αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο μπλοκάρει τα πράγματα και όπως φαίνεται δεν είναι σε θέση για, να λάβει μια απόφαση για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση απόψε προς το Συμβουλίο να λάβει επιτελούς θέση και να ε, εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Κυρία Φόλα, τα ακολουθεί για δύο λεπτά ο συνάδελφος κύριος Ντούραν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεύτσοβιτς, είμαστε μεταξύ μας, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Και ούτως θα πράξουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να δώσει αυτό το κείμενο η Επιτροπή είναι διότι βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος μεταξύ του Συμβουλίου και των μεγάλων επιχειρήσεων που λένε ότι κοιτάξτε άμα δεν πάρετε αποφάσεις τότε εμείς θα συνεχίσουμε θα διώξουμε την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε είστε υποχρεωμένοι να αποφασίσετε εκεί όπου το Συμβούλιο αποδεικνύει ότι είναι δειλό τρομακτικά δειλό γιατί εδώ ουσιαστικά μιλάμε, και το είπατε και εσείς και το ξέρουμε όλοι εδώ, καθόμαστε και μιλάμε για την υγεία 500 εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων καταναλωτών. Αναφέρομαστε σε χημικά προϊόντα, συζητάμε εδώ για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και το λέω ενώπιον του Κοινοβουλίου, του οποίου είμαι μέλος, όπου είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να κάνουμε κάποια πράγματα. Ε, ξέρετε, είναι όλο και περισσότερες οι περιπτώσεις αυτές, διότι ζούμε σε μια κοινωνία όλο και πιο περίπλοκη. Και μας ζητάνε να αποφασίζουμε με διαδικασία κατεπήγοντος, λέγοντας ναι ή όχι. Δεν είναι πια αποδεκτό αυτό. Είναι αδύνατον. Κύριε Σεύτσοβιτς, ε, σας ακούω και θέλω να μάθω. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι προτεραιότητα για τη δημοκρατία, για τους πολίτες. Δεν μπορούμε τώρα να μπαίνουμε μόνο σε λεπτομέρειες του διαδικαστικές. Το να επιβραβεύουμε αυτούς που δεν ψηφίζουν είναι δείγμα δηλίας. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που είπατε ότι το ζήτημα αυτό παραμένει στην ατζέντα της Κομισιόν για το επόμενο έτος. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να μπορέσει να σας βοηθήσει να προχωρήσετε και ε, δράτω με τις ευκαιρίες και συγχωρέστε με, ε, θέλω να αποτύσω φοροτιμής γιατί στην τελευταία θητεία με τον ε, συναδελφό μου Κόρμπετ ε, στην ΑΦΚΟ κάναμε μια γνωμοδότηση και ήθελα να ε, υπογραμμίσω ότι έκανε πολλή δουλειά ο Ρίτσαρτ σε, σε αυτό το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο και λυπάμαι που βλέπω να φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι από εμάς, από το Κοινοβούλιο μας λόγω των ψεμάτων που έχουν πει οι συμπολίτε του. Ευχαριστούμε κύριε Ντύρα. Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Ρόπε. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, συνάδελφοι, σήμερα το πρωί εδώ στο ημικύκλιο συζητήσαμε για την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και καταλήξαμε στο να συμφωνήσουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει η Ευρώπη να γίνει πιο δημοκρατική και θα πρέπει να αφουγκράζεται περισσότερο τους πολίτες. Η Επιτροπή Συγγνώμη, η διαδικασία της επιτροπολογίας έχει επικριθεί γιατί δεν διακρίνεται από δημοκρατικό χαρακτήρα ούτε από διαφάνεια. Δυστυχώς. τα προβλήματα είναι πάρα πολύ έντονα, οπότε έχουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και έχουν επιπτώσεις άμεσες στο τι τρώμε, στην υγεία μας ε, ή ακόμα και για τα ζώα. Από πλευράς των πρασίνων θέλω να προτρέψω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απασχίσει για μια μεταρρύθμιση τη διαδικασία αυτή. να υπάρχει διαφάνεια στις αποφάσεις και θα πρέπει να περιοριστούν οι αρμοδιότητες των ε, κρατών μελών. Να μην μπορούν να τι τις ευθύνες τους ε, αποφεύγοντα να λάβουν αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρόπε για ένα λεπτό ο συνάδελφος ε, από Σπισέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως οι συνάδελφοι έτσι και εγώ στηρίζω τη μεταρρύθμιση της επιτροπολογίας γιατί είμαι πεπισμένος ότι άπαξ και η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις δεν είναι καλό πολλές από αυτές τις πράξεις να παραμένουν χωρίς ε, θέση από πλευρά των χωρών μελών. Και πρόκειται για τα γενετικά τροποποιημένα, για τα φυτοφάρμακα κλπ. Γίνεται συζήτηση εδώ και χρόνια Αυτά τα θέματα τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε και στην προηγούμενη θητεία. Και εδώ πρόκειται για κάτι αρκετά τεχνικό που θα έπρεπε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάπως πιο ενεργά να πιέσει το Συμβούλιο. Ή ίσως να αποφασιστεί κατά πόσο μπορεί να δεχτεί μια αλλαγή το Συμβούλιο. Η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Οπότε φροντίστε παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Ποσπισίλ για ένα λεπτό ο συνάδελφος Χόισεκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτς, η επιτροπολογία είναι ένα από τα φοβερά πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κανένας δεν καταλαβαίνει. Ναι, εμείς. Το κοινό Λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στους πολίτες. Ε, Έπειτα μιλάμε για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία. Και αυτό είναι που λείπει από τη διαδικασία. Τα φυτοφάρμακα ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στη συζήτηση για την επιτροπολογία. Δεν ξέρουν, ε, ο κόσμος δεν ξέρει πώς αποφασίζουν οι χώρες μέλη και λένε οι Βρυξέλλες αποφασίζουν, οι Βρυξέλλες διατάσσουν αλλά τελικά είναι συγκεκριμένες χώρες μέλη, συγκεκριμένες κυβερνήσεις που αποφασίζουν χωρίς να υπάρχει έλεγχος από το κοινό. Και εδώ αυτό πρέπει να αλλάξει. Και χαίρομαι που βλέπω ότι παραμένει η πρόταση της Επιτροπής. Αυτό όμως που τώρα χρειάζεται είναι να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα. Και εδώ όλα να υπάρξουν και νέε πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ελπίζω να επεξεργαστούμε κάποια στιγμή και κυρίως το Συμβούλιο και να πιέσουν και οι πολίτες βέβαια από τη δική τους την πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χόισικ. Για ένα λεπτό η κυρία Μελχιόρ. Thank you very much. I'll be speaking in Danish. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Ε, για τα όσα μόλις είπε ο συνάδελφος, ε, συνεχίζοντας και εγώ, θα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ένωση Ευρωπαίων και βρισκόμαστε εδώ σήμερα διότι οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να μας βάλουν εδώ. Αλλά ξέρω επίσης ότι πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν την Ευρώπη ως κάτι πολύ απόμακρο. Δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά πώς γίνονται τα πράγματα εδώ. Θεωρούν ότι είναι μόνο γραφειοκράτες και τεχνοκράτες. Πολλοί κόσμοι στην Ευρώπη δεν καταλαβαίνει τι θα πει η επιτροπολογία και στην Ευρώπη και εδώ μέσα. Αν δεν μπορέσουμε να εξηγήσουμε την επιτροπολογία, πώς θα μπορέσουμε να θέλουμε να απαιτούμε από τους συμπολίτε μας να καταλάβουν την επιτροπολογία και τι αφορά. Αν δεν μπορέσουμε να εξηγήσουμε την νομοθετική μας διαδικασία στους πολίτες μας, δεν τηρούμε τις βασικές μας αρχές αυτέ που χρησιμοποιήθηκαν για να οικοδομήσουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξηγήσουμε αυτέ τι διαδικασίε στου Ευρωπαίου πολίτε. Γι' αυτό το λόγο, εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση του Renew Europe να μεταρρυθμιστούν οι Γενικέ Αρχέ τη Επιτροπολογία. Και χαίρομαι, κύριε Σεφκοβίτ, που βλέπω ότι και εσεί υποστηρίζετε την ίδια πρόταση. Ευχαριστούμε, κυρία Μέλχιορ. Δεν έχει εγγραφεί κανεί για το Eye, οπότε για να κλείσουμε. Α. Αυτό δεν το είχα προβλέψει. Λοιπόν, κάτι εξαίρεση ο κύριος Κόρμπετ για ένα λεπτό. Όλες. Άκουσα αυτά που είπε η κυρία Μέλκιορ και άλλοι και έχουν δίκιο. Το σύστημα της επιτροπολογίας είναι ένα σύστημα που δεν καταλαβαίνει το ευρύ κοινό. Έχουμε όμως και ένα άλλο σύστημα για εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι κατά εξουσιοδότηση πράξης, που είναι σαφές αυτό το σύστημα. Εξουσιοδοτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποια πράγματα, αλλά αν δεν μας αρέσει αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να το σταματήσουμε και μπορούμε και να αποσύρουμε τις εξουσίες αυτές με τις οποίες έχουμε εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι αυτό ένα επιχείρημα ώστε να χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο τις κατεξουσιοδότηση πράξεις αντί για τις εκτελεστικές. Ο κύριος Σάιρ και εγώ ήμασταν ε, συνεισηγητές για την οριοθέτηση μεταξύ των ε, δύο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο τις κατεξουδότηση πράξεις που είναι πιο δημοκρατικές και διέπονται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστούμε κύριε Κόρμπετ. Ε, εδώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία CatchDI, οπότε δίνουμε στο τέλος για να κλείσουμε το λόγο στον Επίτροπο κ. Σεύτσοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές για αυτή την θετική φιλική ατμόσφαιρα στη συζήτησή μας που έχει τόσο έντονο νομικό χαρακτήρα αυτό το τόσο συναρπαστικό θέμα όπως είπε και ο κύριος Χόισεκ αλλά και Κάρν Μελχιώτη δύσκολα κανείς να εξηγήσει τον κόσμο πώς εφαρμόζονται εφαρμοστικές πράξεις αλλά και πώς εγκρίνονται. Σας διαβεβαιώ, όλα όσα είπατε τα λαμβάνω υπόψη, όλες αυτές τις προτάσεις. Διευκρινίζω ότι και η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν και ο Μιλών υποσχόμαστε όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε και να κάνουμε μεταρρυθμίσεις παντού. Να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη απόδοση ευθυνών για τα θέματα αυτά. Ό,τι είπε ο κύριος Σάιρο, ο κύριος Ροπέ, ο κύριος Ντυρό, όλα όλα αυτά τα σημειώσαμε. Ήταν ξεκάθαρα τα όσα είπατε. Κύριε Κορμπέτ, επίση ευχαριστούμε. Ε, είναι δύσκολο, είμαστε στριμωγμένοι. Όταν κανεί θέλει να υλοποιήσει εφαρμοστική πράξη, κάνει ό,τι θέλει ο συνωμοθέτη. Εσεί. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε και κάποια νομοθετική πράξη. Άρα περιθώριο ελιγμών είναι πολύ μικρό που έχουμε. Οπότε, τέλος πάντων, προσπαθώ να προωθήσω το θέμα, να συνεργαστώ και με το Συμβούλιο και με εσά και πραγματικά να εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες για το μέλλον και να είναι και πιο εύληπτες. Οπότε, σας διαβεβαιωμάστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και η πρότασή μας, στην ίδια ρότα με σας δείχνει και πηγαίνει. Να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο, με την Κροατική και τη Γερμανική Προεδρία, αν χρειαστεί. Και να προωθήσουμε το θέμα. Είναι κρυστάλλινη θέση σας, ε, μια σειρά επιτροπών σας έχουν τοποθετηθεί. Ε, και η Γιούρη και το Κοινοβούλιο. Όσο πιο ξεκάθαρα τοποθετήσετε, τόσο πιο ισχυρός και γνωμεγό όταν συνομιλώ με το, με το Συμβούλιο ότι δηλαδή είμαι στην ίδια γραμμή με το Κοινοβούλιο, οπότε έτσι θα τα πάω καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας, για τις προτάσεις σας, για αυτό το σημαντικό θέμα. Στενά θα συνεργαστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε Σεύτσοβιτς. Κύριε Σεύτσοβιτς. Θα ήθελα αυτή την ε, φιλική ατμόσφαιρα να μην την υπερβάλλουμε με τις ε, εκτελεστικές πράξεις ε, εκπληρώνεται τη βούληση του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν εδώ κάνετε εκτελεστική πράξη ή ερμηνευτική πράξη με αυτά που είπατε. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Σε κάθε περίπτωση ε, ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 16 Ιανουαρίου από τις 9 μέχρι ε, το απόγευμα και μπορείτε να παρακολουθήσετε την Ολομέλεια στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που έμειναν τόσο αργά. Ε, τερματισμός της ε, Ολομέλειας για απόψε.